Καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, μία σημαντική πληροφορία. Επειδή η Επιτροπή Σούρε ψηφίζει την έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προπτικές αύριο, 25 Μαΐου, αποφασίσαμε να ε, κάνουμε τη συνεδρίαση αύριο το απόγευμα στις 2 ακριβώς. Γεγονός που θα επιτρέψει στα μέλη της Επιτροπής μας που συμμετέχουν και στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ να είναι ε, παρόντα και στις δύο ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την αυριανή συνεδρίαση στις 2 το απόγευμα με την ψηφοφορία για την έκθεση DES. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η αλλαγή σας έχει ήδη διαβιβαστεί από, το, από τη γραμματεία την ε, προηγούμενη εβδομάδα και αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με τη συγκεκριμένη τροποποίηση. Έχετε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Να εγκρίνουμε τώρα τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 28ης Μαρτίου και της 4ης Απριλίου. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις πριν από τη λήξη της συνεδρίασης θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω webstream. Να περάσουμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 4. Εντολή για τον τριμερό διάλογο σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012. Συντάκτης της γνωμοδότησης ο Λουίς Μανουέλ Κάπουλας Σάντος, ε, επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή Προπολογισμού. Έχετε όλοι τις κάρτες ε, ψηφοφορίας σας. Έτοιμοι λοιπόν. Καταρχάς, Λουίς θέλεις το λόγο. Όχι. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν απευθείας στην ψηφοφορία. Η ψηφοφορία αφορά την εντολή για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012, για τον οποίο παρουσιάστηκαν 22 τροπολογίες. Κάποιες εξ αυτών θέλουν να καθορίσουν ή να επεκτείνουν τα πιλωτικά προγράμματα. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στην ψηφοφορία. knows Καλώς. Ξεκινάμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 1. Ψήφισαν όλοι. Όχι. Δεν είχε ψηφίσει ο εισηγητής. Είναι δυνατόν. Πέρασε τη ψηφοφορίας. Περιμένουμε λίγο. Πέρασε λοιπόν της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Votato tutti. Ψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 6. 6. Τροπολογία υπαριθμών 6. Οι 4 και οι 5 έχουν καταπέσει. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Επειδή απορρίφθηκε η τροπολογία 3, ψηφίσουμε την τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 4. Πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται και η τροπολογία υπαριθμών 4. Ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία Ντελάνζ, θέλετε το λόγο. Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η τροπολογία υπαριθμών 5 θέλει τη διαγραφή όλων των παραδειγμάτων των τομέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίε, όπω για παράδειγμα το τομέα του ελαιολάδου, γιατί υπάρχουν και άλλοι τομεί οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Τώρα, αντί να τη διαγράψουμε, που ήταν αρχική μου πρόταση, ο να διαγράψουμε τον τομέα του ελαιολάδου για παράδειγμα, καλύτερο θα ήταν να δώσουμε παραδείγματα και από άλλους τομείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Προτείνω λοιπόν να κρατήσουμε τον τομέα του ελαιολάδου και να προσθέσουμε και άλλους τομείς. Ευχαριστούμε την κυρία Ντελάνζ. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 5 λοιπόν. Πέρασε τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία. Ωραία. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 6. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία τη τροπολογία 6. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 7. Πέρασε τη ψηφοφορία για την τροπολογία 7. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία για την τροπολογία 8. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 9. πέρασε ψηφοφορία. ψηφοφορία Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 10. Πέραση τη ψηφοφορίας για την τροπολογία 10. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία για την 11. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 13. Πέρασε η ψηφοφορία για τη 13. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 14. Πέρασε τη ψηφοφορία. Τροπολογία 14 απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 15. Πέραση ψηφοφορίας. Τροπολογία 15 απορρίπτεται. Άρχεται η τροπολογία για το 16. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία για τη 16. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 17. Πέρασε ψηφοφορία για τη 17. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμό 18. Πέρασε τη ψηφοφορία για την 18. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 19. Πέρασε ψηφοφορίας ψηφοφορία για τη 19. Τροπολογία 19 απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορία. η τροπολογία 20 απορρίπτεται. Τροπολογία 21, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 21. Πέραση της ψηφοφορία. εγκρίνεται. Τροπολογία 22 τώρα, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 22. Πέραση τη ψηφοφορία για την 22, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον το συντάκτη. Bene. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5. Έχουμε μία ψηφοφορία πριν περάσουμε στο σημείο 5. Να περάσουμε στο σημείο 5 τώρα. Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευση και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. Συντάκτη τη νομοδότηση ε, Τζάμπα Σαντόρτα Μπάτζη, ε, επί τη ουσία αρμόδια επιτροπή ΙΝΤΑ να ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ε, του κυρίου Ταμπάτζη για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας για την προστασία των ονομασών προέλευσης και τι γεωγραφικές ενδείξει. Η συμφωνία έχει ήδη αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση. Ο κύριο Ταμπάτζη ζητά την, από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του επί του θέματο, να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, μία ψηφοφορία έχουμε μόνο. Πέρασε τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Perfetto. Onorevole... Τέλεια. Κύριε Ταμπάτζη, θέλετε το λόγο? Όχι. Προχωρούμε. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για το σημείο 6. Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα. Συντάκτης ο, κυρία, ο κύριος Άσουαρθ. Και εδώ έχει αποσταλεί η συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ έγκριση και ο κύριο Άσφορντ ζητά από την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την ε, θέση αυτή. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και αυτό με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Δυστυχώς όχι ομόφωνο. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 7. Υγεία των μελισσών και προκλήσεις για το μελισσοκομικό τομέα. Εισηγητής ο κύριος Ταμπάτζη. Θα κάνουμε μία ανταλλαγή απόψεων, παρουσία ενός εμπειρογνώμανα. Καλωσορίζουμε τον καθηγητή Νιούμαν λοιπόν. Κατόπιν πρωτοβουλία του εισηγητή μα, του κυρίου Ταμπάτζη, ο καθηγητή Πίτερ Νιούμαν από το Ελβετικό Κέντρο για την Υγεία των Μελισσών έχει προσυκληθεί για να συζητήσει με την Επιτροπή μα για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Το πρόγραμμα ε, που είναι πρόβλεψη των πρόληψη της υγείας των μελισσών, γιατί πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τις απικίες και έχουμε μεγάλες απώλειες απικίαιων μελισσιών και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μετριάσουμε τις συνέπειες ε, σε δύο επίπεδα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ταμπάτζη για μια σύντομη εισαγωγή και κατόπιν θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Νιούμαν να λάβει το λόγο για 10 λεπτά. Παρακαλώ κύριε Ταμπάτζη, έχετε το λόγο. Kedves σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω λοιπόν για το ζήτημα της ε, υγείας των μελισσών. Εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό καθήκον ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε καταρχάς από το Δεκέμβριο του 2010 μία πολύ λεπτομερή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Απρίλιο επίσης του 2011 έκανε μία δήλωση για το ζήτημα αυτό. Σίγουρα οι συνάδελφοι θα θυμούνται ότι ε, πριν από αυτά, πέρυσι δηλαδή τον Νοέμβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για το ζήτημα της υγείας των μελισσών και ο κύριος Δεκάστρο ήταν αυτός ο οποίος το παρουσίασε εξ ονόματος Επιτροπής μας. Όσον αφορά λοιπόν την υγεία των μελισσών, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο στις ανακοινώσεις που έκαναν αναφέρονται στην δραματική κατάσταση της μελισσοκομίας στην Ευρώπη. Στον τομέα της μελισσοκομίας αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε πολύ σημαντικές ε, ζημίες, πολύ, σημαντικό, πολύ σημαντική μείωση των ε, απικιών μελισσών στην Ευρώπη έχουμε καταγράψει και Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο αντίδοτο, μια μέθοδος προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές στον τομέα της μελισσοκομείας, άνθρωποι που κερδίζουν το ψωμί τους μέσω της εργασίας αυτής. Ο τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός, όχι μόνο για τις μέλισσες αυτές καθ' αυτές, αλλά επειδή και οι μέλισσες λειτουργούν ως μεταφορείς της γύρης. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι η μελισσοκομεία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό αγαθό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε για αγαθό και αυτή τη στιγμή μιλάμε για υπηρεσίε που προσφέρουν ουσιαστικά από τι μέλισσε με τη μορφή τη επικονίαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανταγνωρίσουμε τι σημαντικέ αυτέ υπηρεσίε που προσφέρονται από τι υπηρεσίε από τις μέλισσες, με συγχωρείτε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις απικίες μελισσών με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε και για το ζωικό κεφάλαιο σε άλλες κατηγορίες. Οι περισσότεροι μελισσοκόμοι είναι επίσης ερασιτέχνες, δεν είναι επαγγελματίε. Και κάτι άλλο πρέπει να δούμε είναι ότι δεν αρκεί να προστατεύσουμε τις μέλισσες αυτές καθ' αυτές, αλλά πρέπει συνάμα να αντιμετωπίσουμε τις απικίες ως σύνολο. Θα πρέπει και αυτές να τις προστατεύσουμε. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τον πληθυσμό μελισσών. Ήδη έχουν ξεκινήσει διάφορες συζητήσεις για τις βασικές αιτίες του προβλήματος. Θα μπορούσα γρήγορα να σας παρουσιάσω κάποιες από τις αιτίες αυτές. Υπάρχουν κάποια παράσιτα τα παράσιτα εκείνα τα οποία προκαλούν την βαρόαση των μελισσών. Τα παράσιτα αυτά επιτίθενται στις μέλισσες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε τα παράσιτα αυτά. Υπάρχουν 10 συνολικά προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταπολεμηθεί η βαρόαση. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει καταρχάς είναι να γίνει μία επιστημονική έρευνα προκειμένου να καταλήξουμε σε νέα φάρμακα παρασιτοκτόνα, προκειμένου να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τους παθογόνους αυτούς οργανισμούς που προκαλούν την παρόαση. Πέρα όμως από τα παράσιτα αυτά θα πρέπει να δούμε και ένα άλλο ζήτημα, τις κλιματικές αλλαγές, καθώς επίσης και την έντονη βιομηχανική καλλιέργεια που έχει και αυτή πολύ επιζήμιες επιπτώσεις στις μέλισσες. Έχουν οδηγήσει αυτοί, ε, αυτές οι μορφές καλλιέργειας σε μείωση της βιοπικιλότητας. Και θα πρέπει επίσης να δούμε και τις επιζήμιες επιπτώσεις που έχουν ε, οι, τα παρασιτοκτόνα, τα, οποία, τα ζανιοκτόνα, τα οποία χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στις εντατικές αυτές ε, βιομηχανικές καλλιέργειες. Κανένα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή δεν έχουν εξετάσει βάθος το ζήτημα της, των τοξικών επιπτώσεων που μπορούν να έχουν ορισμένες ουσίες που περιέχονται στα ζυζανιοκτώνα και που καθιστούν σαστικά τα ζυζανιοκτώνα αποτελεσματικά. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιστημονική έρευνα για τα συστατικά των ζυζανιοκτώνων και για τις τοξικές ενδεχόμενες επιπτώσεις τους και θα πρέπει οι ουσίες αυτές στη συνέχεια να υποκατασταθούν από άλλες ουσίες μη βλαβερές δηλαδή να έχουμε ζυζανιοκτώνα τα οποία να είναι μεν αποτελεσματικά, αλλά να μην είναι επιζήμια για τις μέλισσες. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο απροχώρητο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα ζυζανιοκτώνα. Πρέπει να, κάνουμε, πρέπει να έχουμε μια επιλεκτική στάση απέναντι στι ουσίε αυτέ και να λάβουμε υπόψη μας και την υγεία των μελισσών. Κάτι ακόμα πρέπει να γίνει είναι η, η κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση. 90% των μελισσοκόμων είναι εραστέχνε, όπως είπαμε και δεν έχουν το κατάλληλο επίπεδο επιμόρφωσης κατάρτισης. Αυτό ισχύει στα περισσότερα κράτη-μέλη. Θα μπορούσα να δώσω για παράδειγμα την κατάσταση στην Ουγγαρία. Στα πλαίσια του δικού μας συστήματος προστασίας της υγείας των ζώων, υπάρχουν ορισμένοι που έχουν ε, ειδικευτεί στην υγεία των μελισσών. Ωστόσο, υπάρχουν άλλοι δικοί, άλλοι κτηνίατροι, οι οποίοι δεν είναι δικευμένοι σε ζητήματα υγείας των μελισσών. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Και υπάρχει και ένα στοιχείο στο οποίο θα αναφερθώ. Αν δούμε τώρα το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής, ένα ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι και όλα αυτά τα προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία των μελισσών. Ο μόνος τρόπος για να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά είναι σε κοινοτικό επίπεδο. Σαφώς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μονομένες χώρες και μονομένες περιφέρειες στο πλαίσιο μιας χώρας, δεδομένης όμως της των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μελισσών δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σφαιρικά, διασυνοριακά. Όπω γνωρίζετε, οι μέλισσε μετακινούνται από τη μία περιοχή στην άλλη. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια κοινή ευρωπαϊκή σφαιρική λύση για τα προβλήματα υγεία των μελισσών. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο προσκάλεσα και με τη σύμφωνη γνώμη τη κυρία Λούλινγκ τον Πέτερ Νόμαν, ο οποίο θα μα μιλήσει για το δίκτυο αυτό που ονομάζεται Κολοσσός όπως είπαμε, το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με τη χρησιμοποίηση των ζυζανιοκτώνων, αλλά έχει να κάνει και με το ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα στατιστικά δεδομένα στα χέρια μας. Δεν έχουμε ακόμη και ακριβά στοιχεία για τον αριθμό των μελισσιών. Πρέπει να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει τους ε, μελισσοκόμους και πρέπει να δούμε βέβαια αν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εποπτείας, παρακολούθησης και στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα να είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε πώς εξελίσσονται οι πληθυσμοί μελισσών και πώς η μείωση πολλές φορές των απικιών μελισσών επηρεάζει την μεταφορά της γύρης. Πρέπει επίσης να γίνουν οι απαραίτητες ε, επιστημονικές έρευνες, να μην χρηματοδοτούμε μόνο την παραγωγή φαρμάκων, αλλά και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά καθ' αυτά. Πολλές φορές οι ανακοινώσεις και του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δίνουν κάποιες πρώτες λύσεις, αναφέρουν κάποιες πρώτες ιδέες. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μόνο που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είναι να κάνουμε ένα απολογισμό της κατάστασης και δημιουργούμε απλώς κάποιους καταλόγους με τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή σε μια ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων αυτών. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταμπάτζη. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον εμπειρογνώμονά μας, τον Πίτορ Νιούμεν Έχετε 10 λεπτά το πολύ. Παρακαλώ κύριε Νιούμαν. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα να σας πω ότι οι μέλισσες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τα οικοσυστήματα στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας και δραματίζουν ένα κεντρικό ρόλο επίσης στην ε, ισορροπημένη, σωστή ανθρώπινη διατροφή. Αν τα λάβετε λοιπόν όλα αυτά υπόψη σας, θα δείτε στην διαφάνεια αυτή την οποία μάλλον δεν μπορείτε να δείτε, μια φωτογραφία από μια πικία μελισσών. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές μέλισσες ε, οι οποίες ε, έχουν πεθάνει. Βλέπετε τη φωτογραφία αυτή πως ε, καταδεικνύει πάρα πολύ καλά την μείωση του πληθυσμού των μελισσών. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα όπως η διατροφή, η χρησιμοποίηση των ε, ζυζανιοκτώνων, διάφοροι παθογόνοι παράγοντες, καθώς επίσης ακόμα και η ίδια μελισσοκομεία δημιουργεί ένα άγχος, ένα στρες στις μέλισσες. Υπάρχουν επίσης ε, άλλοι παθογόνοι παράγοντες οι οποίοι συνδέονται με την υγεία των μελισσών όπως η ελονοσία. Επίσης υπάρχουν κάποια ζενοκτώνα τα οποία μπορούν να καταστήσουν τις μέλισσες πιο ευάλωτες στο να αρρωστήσουν από κάποιους παθογόνους παράγοντες. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους και υποδηγούν σε αυτή την πολύ άσχημη κατάσταση για τις μέλισσες. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί πληθυσμοί μελισσών οι οποίες επηρεάζονται από τα παράσιτα αυτά που προκαλούν την βαρόαση των μελισσών. Πολλές φορές βέβαια με την έκθεση στα ζανιοκτώνα και με τους παθογόνους παράγοντας δεν ξέρουμε ακριβώς πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Επίσης μας λείπει η γνώση για ορισμένους παθογόνους παράγοντες καταλαβαίνετε ότι οι μέλισσες αντιδρούν πολύ διαφορετικά από ότι τα ζωικά κεφάλαια σε, άλλη, σε άλλα είδη. Επίσης είναι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει χρηματοδοτηθεί αρκετά, δεν έχουν γίνει απαραίτητες έρευνες και δεν γνωρίζουμε επομένω ποια είναι τα παράσιτα αυτά τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τις μέλισσες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει πλέον το απαραίτητο επίπεδο συνεργασίας προκειμένου να καταφέρουμε να αποκομίσουμε τη γνώση αυτή που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Βλέπετε εδώ πέρα πώς λειτουργεί το δίκτυο αυτό, το οποίο έχει το όνομα Κόλοσσος. Έχουμε 269 μέλη από 55 χώρες. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, η πρόκληση είναι ιδιαίτερα μεγάλη για μένα για να καταφέρουν διαχειριστώ το δίκτυο αυτό. Έχουμε μια πολύ καλή κάλυψη στην Ευρώπη και παρουσία επίσης στη Βόρεια και Νότια Αμερική, καθώς επίσης και στην Αφρική και την Ασία. Μέσω των διαφορετικών αντένων που έχουμε και των διαφορετικών ομάδων εργασίας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά ζητήματα τα οποία βάλουν την υγεία των μελισσών. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τα απαραίτητα πρότυπα, τι απαραίτητε προδιαγραφέ για την παρακολούθηση και την εποπτεία τη υγεία των μελισσών, κάτι το οποίο πουσιάζει αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να εντοπίσουμε παράγοντε οι οποίοι οδηγούν σε πολύ σημαντική μείωση του πληθυσμού των μελισσών και θέλουμε επίσης να δημιουργήσουμε και τα απαραίτητα μέτρα έκτακτης ανάγκης καθώς επίσης και στρατηγικής ε, προστασίας της υγείας των μελιτών. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να καταφέρουμε να συλλέξουμε αξιόπιστα δεδομένα για την μείωση των απικιών μελισσών. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το πρόγραμμα ε, προστασίας του περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ισχύει σε 30 χώρες και βέβαια και στην Κίνα και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ένα άλλο μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε B-Book, ένα εγχειρίδιο για τις μέλισσες. Εδώ πέρα προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε κάποιες μεθόδους, τυποποιημένες και αυτές, προκειμένου να αναλύσουμε καλύτερα την κατάσταση της υγείας των μελιτών, μελισσών σε διάφορες απικίες. Έχουμε επίσης δύο προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται BDOC και έχει ως στόχο την συλλογή πληροφοριών για τους παθογόνους παράγοντες που βάλουν κατά των μελισσών και ένα ακόμα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται STEP το οποίο καταγράφει το γενικότερο καθεστώς καθώς επίσης και στις τάσεις όσον αφορά τα έντομα επικονιαστές στην Ευρώπη. Το πρόβλημα βέβαια που έχουμε είναι ότι η χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμη. Ακόμα και αν υπάρχει μία βραχυπρόθεσμη και μέσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, δεν αρκεί προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα σημαντικά προβλήματα που έχουμε. Δεν μπορούμε μέσα σε τρία-τέσσερα χρόνια να διορθώσουμε όλα αυτά τα οποία δεν γίνανε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που δεν υπήρχε χρηματοδότηση και έρευνα για την μελισσοκομεία. Όλα λοιπόν τα προγράμματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την έρευνα και τη διάσωση των μελισσών ποιε είναι οι γενικότερε προκλήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή για τη μελισσοκομία. Βλέπουμε ότι γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνονται οι απικίες μελισσών, μειώνονται επίσης και οι μελισσοκόμοι. Έχουμε όλο και περισσότερα παράσιτα τα οποία καθιστούν τη μελισσοκομία έναν τομέα ο οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ απικίε μελισσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν μολυνθεί και αν δεν καταφέρουμε να βοηθήσουμε του μελισσοκόμου, μέσα σε δύο-τρία χρόνια θα καταστραφούν πάρα πολλέ απικίε. Καταβάλλονται λοιπόν πάρα πολύ σημαντικέ προσπάθειε και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε μια βιώσιμη κατάσταση. Δεν έχουμε μια βιώσιμη λύση και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πόσε λίγε γνώσει έχουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης βλέπουμε ότι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν σημαντικές εισαγωγές πληθυσμών μελισσών όπου υπάρχουν από χώρε όπως η Αυστραλία, όπου υπάρχουν σημαντικοί υγειονομικοί κίνδυνοι για τους πληθυσμούς των μελισσών. Πολλές φορές δηλαδή μαζί με τους πληθυσμούς αυτούς φτάνουν και επικίνδυνα παράσιτα. Δεν έχουμε απαραίτητε γνώσει λοιπόν όσον αφορά την υγεία των μελισσών, δεν έχουμε την απαραίτητη κατάρτιση όσον αφορά του εμπλεκόμενου στον μελισσοκομικό τομέα. Όπω είπαν, περισσότεροι μελισσοκόμοι είναι αεραστεχνέ, το κάνουν αυτό στον ελεύθερο χρόνο του. Σαφώ οι άνθρωποι αυτοί ε, παρέχουν πολύ σημαντικέ υπηρεσίε επικονίαση και δεν λαμβάνουν την απαραίτητη αναγνώριση από τα κράτη-μέλη. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στην κατάσταση από τη μία χώρα στην άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετική κατάρτιση, διαφορετική υποδομή, διαφορετικές μέθοδοι ελέγχου της ποιότητας. Ποιοι είναι οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στο μελισσοκομικό τομέα. Σαφώ στο κέντρο έχουμε του μελισσοκόμου. Έχουμε όμω ε, διάφορου επιστήμονε ειδικευμένου στι μέλισσε. Έχουμε τον, την ίδια τη βιομηχανία, του κτηνιάτρου. Πιστεύω ότι η βιώσιμη λύση μπορεί να έρθει μόνο με την ε, βοήθεια και τη συμμετοχή της βιομηχανίας. Επιτέχουμε τις κυβερνήσεις. και τους ηθήνοντες για την ε, χάραξη πολιτικής. Τις είναι οι λύσει τώρα που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Καλύτερη κατάρτιση, καλύτερη ευαισθητοποίηση για όλους του εμπλεκόμενου παράγοντες, αυξημένη γνώση για τις υπηρεσίε επικονίασης, κάποιες συντονισμένες προσεγγίσεις οι οποίες θα συντονίζουν όλους τους εμπλεκόμενους προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη λύση, ποια είναι τα απαραίτητα μέσα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Λιγότερες εισαγωγές μελισσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε επίσης ένα καλό σύστημα networking, δηλαδή το σύστημα αυτό, το δίκτυο κολοσσός. Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα ότι δημιουργήθηκε επιτέλους ένα εργαστήριο αναφοράς και θα πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν με το εργαστήριο αυτό προκειμένου να γίνουν συντονισμένες ερευνητικές ε, ε, προσπάθειες χωρίς να υπάρχει επικάλυψη προσπαθειών. Επίσης, χρειαζόμαστε μια βελτιωμένη κατάρτιση όλων των εμπλεκομένων και τέλος περισσότερη και πιο βιώσιμη έρευνα για τις μέλισσες. Προκειμένου να καταπολεμήσουμε την βαρόαση, χρειαζόμαστε πολλά έτη έρευνας και χρηματοδότησης έρευνας αυτής. Θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των λύσεων που προτείνω. Χρειαζόμαστε πιο συστηματική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω όσον αφορά τη χρηματοδότηση τη έρευνα, προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που πλήττουν τον παράγοντα τη μελισσοκομ... μελισσοκομία. Θα ήθελα εδώ πέρα να σας να ευχαριστήσω το δίκτυο κολοσσός όλους τους εμπλεκόμενους στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Πίτερ Νόιμαν. Ε, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Ταραμπέλα καταρχάς και μετά ο Τζέιμς Λίγκολσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα τον πραγματογνώμονα με μεγάλη προσοχή γιατί πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια και το οποίο φαίνεται ότι δεν εξαλείφεται εύκολα. Όντως χρειάζονται μέσα. Καθορίζουμε το πρόβλημα. Άκουσα τον εμπειρογνώμονα που μίλησε μιλήσε για την μείωση του αριθμού των μελισσών που έχει ξεκινήσει από το 85 και ότι όταν εξαφανιστούν οι μέλισσες θα εξαφανιστεί και η ανθρώπινη ζωή. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε αντικειμενικοί και ας προσπαθήσουν οι επιστήμονες να μας πούν πού είναι το πρόβλημα. Ακούμε ότι φταίει κάποιος και κατόπιν η αιτία είναι διαφορετική και δεν πρέπει εδώ να κατακαιρματίσουμε τα μέσα που διαθέτουμε και τις προσπάθειες μεταξύ των επιστημόνων και των δίθεν επιστημόνων, οι οποίοι όντως εργάζονται για την προάσπιση διαφορετικών ε, συμφερόντων, διαπιστώνουμε ότι και η βαρόαση των μελισσών, αλλά και άλλες ασθένειες θα πρέπει να εξαλειφθούν. Από την άλλη μεριά ακούμε ότι τα ζυζανιοκτώνα και τα παρασιτοκτώνα επιδεινώνουν πολλές φορές την κατάσταση. Ας επικεντρωθούμε όμως στην έρευνα γιατί εδώ φαίνεται ότι χρηματοδοτούμε κάποιες μελέτες χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα. Όντως λοιπόν πρέπει να αυξήσουμε και τα μέσα και τις προσπάθειές μας στα πλαίσια της κοινή αγροτικής πολιτικής. Πρόκειται για το μέλλον της βιοποικιλότητας. Αλλά έχω λίγο κουραστεί γιατί ακούω διαφορετικούς εμπειρογνώμονες να κάνουν διαφορετικές προτάσεις. Να αναλύσουμε τους διάφορους παράγοντες, παθογόνους και άλλους και ας μας προταθεί μία λύση, μία πρόταση ε, ή κάποιες συμβουλές. Εδώ και 25 χρόνια μελετάμε και λύση δεν υπάρχει. Δεν ξέρω σε πόσα χρόνια κάτι θα γίνει. Ας δώσουμε ένα χρονικό διάστημα 10 ετών, ας σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε κάποιους ερευνητές και κάποια λόμπι γιατί χάνουμε το χρόνο μας και σπαταλούμε και δημόσιο χρήμα. Δεν είμαι επιστήμονας, αλλά θα ήθελα οι επιστήμονες κάπως να συμφωνήσουν ως προς τη μέθοδο εργασίας. Αν δεν μπορούν να το κάνουν, ας δοκιμάσουμε τη μία μέθοδο και αν δεν έχουμε αποτέλεσμα, ας στραφούμε προς μία άλλη. Γιατί κινδυνεύουμε σε κάποια χρόνια να μην υπάρχει πλέον ούτε μία μέλισσα και καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύουμε να βρεθούμε μπροστά σε ένα πιο σοβαρό πρόβλημα. Οι ερευνητές ψάχνουν, ερευνούν, ας βρουν και κάτι επιτέλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. James Nicholson και μετά ο κύριος Νικουλέσκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας απασχολεί. Η κυρία Λούλινγκ ήταν ε, στην πρωτοπορία και είχαμε στηρίξει τις προσπάθειές της να βρούμε κάποιες λύσεις για αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο. Δεν είναι θέμα που μας απασχολεί εδώ και ένα ή δύο χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και όλοι οι τομείς πλήττονται από το φαινόμενο αυτό. Περισσότερα χρήματα, περισσότερες προσπάθειες μας ζητούν σήμερα, περισσότερες ε, κλινικές ε, έρευνες για να εντοπιστούν οι πραγματικές αιτίες του φαινομένου αυτού. Δεν έχουν βρεθεί ακόμα 100%. Σήμερα συνεχίζουν να πεθαίνουν οι μέλισσες, να μειώνεται ο αριθμός τους και σαφώς και θα πρέπει να υλοποιηθούν κάποια από αυτά που έχουν ε, ερευνηθεί μέχρι τώρα. Εγώ είμαι από την Ιρλανδία και βεβαίως στην περιοχή μου υπάρχουν όλα αυτά τα φαινόμενα που περιγράψατε. Ακούσαμε ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες, περισσότερα χρήματα, αλλιώς δεν θα υπάρχουν πλέον μέλισσες σε λίγα χρόνια. Όπως είπε και ο Μάρκ Ταραμπέλα, δεν είμαι ούτε εγώ ειδικό, δεν είμαι επιστήμονας. Αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τι δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Υπάρχει κάτι το οποίο και ερωτώ τον ειδικό μας. Υπάρχει κάτι που έχει εντοπιστεί και θα έπρεπε να είχαμε κάνει και δεν το κάναμε. Νομίζω αυτό προσπάθησε να ρωτήσει και ο Μάρκ. Τόσα χρόνια επανέρχεται το πρόβλημα αυτό και θα πρέπει ίσως να αναρωτηθούμε τι θα μπορούσε να είχε γίνει, πώς θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα στις ερευνές μας για το ποια είναι η αιτία αυτού του αφανισμού. Τι να σας πω, μπορούμε να πούμε ότι δεν φταίμε εμείς που η έκρηξη του εφεστίου γέμισε την ατμόσφαιρα με τέφρα. Αλλά όσον αφορά τον αφανισμό των μελισσών, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια συγκεκριμένη αιτία. Θα πρέπει κάποια στιγμή να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Κύριος Νικολέσκο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, προσκεκλημένο μας. Και εγώ δεν είμαι ειδικό στις μέλισσες, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις παρόλα αυτά. Η μελισσοκομεία μπορεί να είναι χόμπι για παθιασμένους ερασιτέχνες. Η εξαφάνιση όμως ολόκληρων απικιών μελισσών είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε όλοι. Εδώ βεβαίως και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όλους τους μελισσοκόμους να συνεχίσουν αυτή τη δραστηριότητα επαγγελματική ή ερασιτεχνική. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον ειδικό. Υπάρχουν κάποιες απικίες μελισσών, κάποια είδη μελισσών, κάποιες ράτσες που είναι πιο ανθεκτικές. Επίσης, τι έχουμε να πούμε όσον αφορά τα εντομοκτώνα. Υπάρχουν ίχνη και στο μέλι. Ευχαριστώ, κυρία Ρέιμερ. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, όλοι συμφωνούμε στην Επιτροπή ότι πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα. Η υγεία των μελισσών μας απασχολεί. Επίσης έχουμε σημαντικά προβλήματα και με όλους αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν την δραστηριότητα των μελισσοκόμων όταν αυτοί σταματήσουν. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και αυτό βεβαίως είναι ένας από τους λόγους που μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των μελισσών. Χρειάζονται βεβαίως χρήματα μέσα και συντονισμός. Ο συντονισμός είναι η δουλειά η δική μας, των πολιτικών. Δηλαδή τα μέσα που διαθέτουμε να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο. Το πρόγραμμα αυτό το παγκόσμιο, το οποίο έχει σαν σκοπό τον συντονισμό, θα πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια συγκρίσιμα αποτελέσματα. Ή ο καθένας θα κάνει την ε, δουλειά του χωρίς να μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. Αυτό είναι μια ερώτηση που σας κάνω. Δεύτερον, θα ήθελα να ξέρω εάν οι ερευνητέ ανταλλάσσουν στοιχεία και πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσουμε και εδώ να εξοικονομήσουμε κάποια μέσα. Αν δηλαδή στην κάθε χώρα υπάρχουν μονάδες ερευνητών, ομάδες που εργάζονται, θα μπορούσαμε ίσως να αποφύγουμε διπλή εργασία και κατασπατάληση μέσων και κονδυλίων εάν υπήρξε συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ερευνητών. Έχουμε περιορισμένα μέσα, γι' αυτό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε εν ώψη της οικονομικής κρίσης να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στο πώς δαπανώνται αυτά τα κονδύλια. Κυρία Μαγκίνης και μετά ο Μάρτιν Όσλιχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συμφωνήσω και εγώ με τα σχόλια των συναδέλφων και να πω ότι θα πρέπει να μας ενδιαφέρει η έρευνα που είναι στοχευμένη και έχει αποτελέσματα. Αλλά εγώ νομίζω ότι έχουμε και ένα προβληματισμό ευρύτερο από τη συζήτηση αυτή. Έχουμε τις μέλισσες οι οποίες ε, ε, είναι αντικείμενο μελισσοκομεία, αλλά υπάρχουν και άλλε μέλισσε οι οποίε κυκλοφορούν ελεύθερε. Δεν άκουσα κανένα να συζητά την υγεία των άγριων μελισσών και τη συνεισφορά τους ε, στην επικονίαση και τη βιοπικιλότητα μπορεί οι εμπειρογνώμονες να μπορούν να θίξουν και αυτά τα θέματα, διότι νομίζω ότι και αυτά μας απασχολούν. Και να πω επίσης ότι το γεγονός ότι υπάρχουν ερασιτέχνες στον κλάδο αυτό είναι μάλλον και τμήμα του προβλήματος. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτό και θα πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο το θέμα από ευρύτερη σκοπιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρτινόλσεν και μετά η κυρία Έρανς Καρθία. Το πρόβλημα είναι ότι στην ε, Ευρώπη δεν είναι εύκολο να κανείς ε, ερασιτέχνης με Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να βρει κάποιος να τον διαδεχθεί, να αναλάβει τη δραστηριότητα αυτή μετά Χρειάζεται λοιπόν εδώ να κάνουμε μια συγκεκριμένη προσπάθεια όσον αφορά την κατάρτιση των μελισσοκόμων. Και είναι παλιό το πρόβλημα, το γνωρίζουμε. Έρευνα έχει γίνει, μελέτες έχουν γίνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των ε, μελετητών. Το θέμα της βαρόασης είχαμε ακούσει ότι είναι ένα πρόβλημα μεταξύ πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μέλισσες. Ότι χρησιμοποιούνται δηλαδή πολλές χημικές ουσίες στη Γεωργία. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε στη Νότια Γερμανία ε, το θέμα της ε, αντιμετώπισης ασθενειών και ζυζανιοκτώνων για το καλαμπόκι, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να εξαφανιστούν ολόκληρες απικίες μελισσών. Το ίδιο έγινε και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για κάποια λουλούδια. Βεβαίως και χρειαζόμαστε μια πιο πράσινη και προσεκτική γεωργία, αλλά χρειαζόμαστε και μια πιο πολύχρωμη, όχι μόνο πράσινη αγροτική πολιτική. Δηλαδή είναι απαραίτητο να προσέξουμε ιδιαίτερα την ε, ποικιλομορφία, έτσι ώστε οι μέλισσες να μην βρεθούν χωρίς τίποτα να φάνε. Ευχαριστούμε κύριε Ραντς Καρσία τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς. Επανειλημμένως είχαμε τη δυνατότητα όταν πήγαμε και στη Ρουμανία να ακούσουμε κάποιον μελισσοκόμο ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για την κατάσταση της μελισσοκομίας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τους ελέγχους και την εποπτεία που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη για να ε, ελέγξουμε για ποιο λόγο αυξάνεται η θνησιμότητα των μελισσών, αλλά θα ήθελα να ακούσω και κάποια πράγματα για τα κλιματοϊκά φαινόμενα και επίσης για το κατά πόσον η απώλεια βιοποικιλότητας που έχουμε ήδη στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο επηρεάζει τη ζωή των μελισσών και την ε, επιβίωσή τους. Άκουσα ήδη κάποιους εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με το θέμα στην Ισπανία, οι οποίοι ερευνούν το θέμα και μιλούσαν για τη θνησιμότητα που παράγεται από τη χρήση και τον πολλαπλασιασμό της χρήσης των κινητών ε, τηλεφώνων και φαίνεται ότι έχουν αναπτύξει μεταξύ τους ακόμα και μία γλώσσα ε, για να στέλνουν ένα σήμα κινδύνου όταν είναι κοντά σε λήψη κινητής τηλεφωνίας. Ε, φαίνεται ότι τους επηρεάζουν όλα τα προβλήματα που ε, προκύπτουν και για μας από την κινητή τηλεφωνία. Θα θέλαμε λοιπόν όταν συνεργαζόμαστε να συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες που θα έχουν μελετήσει καλά τα θέματα και με τεχνικούς που θα γνωρίζουν τα πράγματα και τα τεχνικά στοιχεία για να μπορούμε να λάβουμε και εμείς μία πληροφορημένη απόφαση. Δεν μ' αρέσει να ακούω ότι επικρίνονται, για παράδειγμα, μόνο οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί και άλλες επικρίσεις όταν δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη, κανένα σοβαρό επιστημονικό στοιχείο που να καταδεικνύει ότι ε, επιδεινώνεται η κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα φάρμακα για να επιτεθούμε σε όλες τις ασθάνειες που τις πλήττουν και η χρήση των αντιβιωτικών και το τι συνέπειες μπορεί να έχουν είναι κάτι ενδιαφέρον. Αλλά επαναλαμβάνω, πάντα θα πρέπει να βασόμαστε σε απτά επιστημονικά στοιχεία και όχι ε, να μένουμε σε προκαταλήψεις ε, με συγκεκριμένες ιδέες για να διαμορφώνουμε άποψη. Ολοκληρώνοντας, η κυρία Λούλινγκ. Παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη μου στην Νομισματική Επιτροπή. Γι' αυτό και δεν ήμουν εδώ από την αρχή της συζήτησης. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η συζήτηση με φέρνει πίσω 15 χρόνια. Είναι ευχάριστο στην ηλικία μου αυτό. Είμαι μόνιμη εισηγήτρια για θέματα γεωργικής πολιτικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όλα αυτά που ακούστηκαν, προτάθηκαν, τα έχουμε γράψει και ξαναγράψει και ξαναξαναγράψει σε γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις. Όλα αυτά, όλα αυτά. Εδώ και πολλά χρόνια η Επιτροπή κάνει ότι δεν ακούει. Μετά την πρώτη μου έκθεση είχαμε ζητήσει μάλιστα και ε, ένα ποσό για την επικονίαση για τους Ευρωπαίους αγρότες. Το 1995 το είχαμε ζητήσει αυτό. Σαν αποτέλεσμα, το μόνο που πήραμε το 1997 είναι ένα ποσό για την διάθεση της αγοράς του μελιού αλλά πρέπει να σας πω ότι ξεκινήσαμε με 10 εκατομμύρια και φτάσαμε στο πενιχρό ποσό των 30 δικατομμυρίων ευρώ για την μελισσοκομεία στην Ευρώπη. Το μόνο που καταφέραμε να επιτύχουμε. Και αυτό γιατί βεβαίως υπάρχει το θέμα της συγχρηματοδότησης ε, του ύψους του 50% από το μέρος των κρατών μελών. Είχαμε ζητήσει το θέμα των μελισσών να συμπεριληφθεί στην κτηνιατρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας απάντησαν όχι. Αυτό αφορά μόνο τις ε, ασθένειες που μπορεί να εξαλειφθούν. Φαίνεται δηλαδή ότι οι ασθένειες των μελισσών δεν μπορεί να εξαλειφθούν. Έτσι ε, αντιδράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι λίγο πιο ανοιχτή, έχει δείξει περισσότερη προσοχή, όχι όμως το Συμβούλιο, αλλά σε επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά τα έχουμε πει και ξαναπεί. Ας μην ξαναρχίσουμε από την αρχή η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να ακολουθήσουν επιτέλους τις προτάσεις της ε, Επιτροπής μας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ ξεκίνησα το 1995 και ακολούθησα ουσιαστικά, ήμουν διάδοχος του κυρίου Μπέγκε που είχε κάνει τον ίδιο αγώνα πριν από μένα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μας ακούσει η Επιτροπή. Εδώ και 15 χρόνια λέμε τα ίδια. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε τα ίδια από την αρχή, απλώς να εκτελέσει η Εκτελεστική Επιτροπή. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να διαθέσει τίποτα παραπάνω από 32 εκατομμύρια για να σωθεί η μελισσοκομεία, τότε ας εγκαταλείψουμε τις προσπάθειές μας. Αν είμαστε τόσο φτωχοί και δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ούτε την έρευνα, ούτε όλα αυτά που έχουμε ζητήσει, τότε δεν έχει νόημα να κάνουμε εκθέσεις και ψηφίσματα. Ας μας πει επιτέλους η Επιτροπή αν είναι διατεθειμένη να μας ακολουθήσει και να κάνει κάποια συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, κάτι που έχουμε ζητήσει εδώ και χρόνια, επαναλαμβάνω. Θα ήθελα να πω στον εμπειρογνώμονα, τον οποίο άκουσα με μεγάλη προσοχή, ότι καταρχήν πιστεύω ότι αυτό που είπατε, ότι οι ερασιτέχνες μελισσοκόμοι δεν γνωρίζουν τίποτα, δεν μπορώ να το δεχτώ. Καταρχήν, μόνο το 3% των μελισσοκόμων είναι επαγγελματίες. Μπορείτε να αντικαταστήσετε από τη μία μέρα στην άλλη αυτές τις 500.000 ερασιτέχνες μελισσοκόμους με επαγγελματίες. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά τις ενώσεις μελισσοκόμων στην χώρα μου. Βεβαίως και κάνουν προσπάθεια κατάρτισης. Γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Δεν μπορεί κάποιος να γίνει επαγγελματίας μελισσοκόμος από τη μία μέρα στην άλλη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εμείς να αγνοήσουμε όλους αυτούς τους τέχνες μελισσοκόμους ή να τους υποτιμήσουμε. Στο ψήφισμα που έχουμε υιοθετήσει λέμε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για το σημερινό φαινόμενο. Κάποιοι μιλούν για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Άλλοι μόνον για τα παρασιτοκτόνα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο είναι σωστό. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση και το πρόβλημα είναι η προστασία της βιοποικιλότητας. Το λέμε, το επαναλαμβάνουμε, χρειάζονται μέσα για να πετύχουμε αυτά που ζητάμε στα ψηφίσματά μας, δηλαδή να διασφαλίσουμε δίπλα στις μόνο να υπάρξουν καλλιέργειες διαφορετικές για να μπορέσουν να τραφούν και να επιζήσουν οι μέλισσες. Είναι όπως ακριβώς θα έλεγα και για τις ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορούμε να ζήσουμε αν τρεφόμαστε μόνο με ενός είδους τρόφιμα. Η Εκτελεστική Επιτροπή, επαναλαμβάνω, μας αγνοεί δεν ακούει, τι παραπάνω να ζητήσουμε. Τα έχουμε ζητήσει όλα πια στις προηγούμενες εκθέσεις μας. Εδώ και 15 χρόνια τα ζητάμε. Ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστούμε. Βλέπετε ότι είναι πλήρης υποστήριξη της Επιτροπής για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Και επειδή ετέθησαν μία σειρά από ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ακούσουμε αμέσως τον κύριο Λαντομάντα για τη γνώμη της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου και τον εμπειρογνώμονα που παρενέβησαν με τόσο εύστοχο και ενδιαφέρον τρόπο σε απάντηση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2010. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά που είπε ο εισηγητής για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο καλύτερα θα ήταν να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει έλλειψη στοιχείων και υπάρχει και ανάγκη για απτές λύσεις. Αρκετοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στην ανάγκη αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, καλύτερη συνέργειας μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στη διάρκεια του προηγούμενου έτους όρισε καταρχάς ένα νέο εργαστήριο αναφοράς για την υγεία των ε, μελισσών, το, ε, ένα εργαστήριο στη Γαλλία, το οποίο συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία των μελισσών. Επίσης, ξεκίνησαν κάποια προγράμματα επιμόρφωσης για υπαλλήλους μέσω του προγράμματος Better Training for Safer Food, προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτασης για τους μελισσοκόμους, επίσης περιλαμβάνονται και στα εθνικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται τακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή η χρηματοδότηση στα εθνικά προγράμματα υποστήριξης της μελισσοκομείας αυξήθηκε κατά 25 περίπου 100 για το διάστημα από το 2011 έως 2013 ανέρχονται πλέον στα 32 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί επίσης τρία τουλάχιστον σημαντικά ερευνητικά προγράμματα και το πρόγραμμα Κολοσσός είναι το ένα εξ αυτών, αλλά υπάρχουν και τα προγράμματα BIDOC και STEP, τα οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο τις μελιτοφόρους μέλισσες, αλλά και άλλα έντομα επικονίασης. Αυτό διότι προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που άπτονται όχι μόνο των μελισσών αλλά και άλλων εντόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία της επικονίασης. Κάποιος από τους ομιλητές είπε ποια είναι η πιο σημαντική δράση η οποία θα πρέπει να γίνει. Εξαιρετική ερώτηση, θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποιες απαντήσεις. Είναι δύσκολο να απαντήσουμε με μία και μόνο απάντηση. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει ε, στο εγγύς μέλλον να κάνει τα εξή. Καταρχάς θέλουμε να οργανώσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα επιοπτείας για να παρακολουθούμε τη διάσταση του φαινομένου της νησιμότητας των μελισσών, γιατί αυτή είναι η βασική πτυχή και αυτό θα θέλαμε να το κάνουμε σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Επομένως δεν μιλάμε μόνο για μια επιστημονική πρωτοβουλία, αλλά για κάτι επιπλέον το οποίο θα ε, απαιτεί και τη συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία της εποπτείας. Αυτό θα συζητηθεί σε διάσκεψη στις 6 και 7 Ιουνίου. Στη διάσκεψη αυτή έχουν προσκληθεί όλοι οι εμπειρογνώμονες από τα εθνικά εργαστήρια, τα κρατημέλη και φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ευπρόσδεκτο σε αυτή τη διάσκεψη. Εξετάζουμε επίσης εκ νέου και την νομοθεσία για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη ε, μελισσοκομεία, τα κτηνιατρικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα από τα πρωταρχικά προβλήματα. Αναθεωρείται όλη η νομοθεσία για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της ε, διάθεσης ε, θεραπευτικών προϊόντων κατά των διαφόρων ασθενειών των μελισσών. Ενισχύουμε επίσης τα κριτήρια για την έγκριση φυτοφαρμάκων. Αυτό είναι τμήμα της νέας νομοθεσίας. Αυξάνουμε τη χρηματοδότηση στα ερευνητικά προγράμματα και επανεξετάζουμε τους κανόντες της υγείας των ζώων όσον αφορά τις μέλισσες, των εντόμων σε αυτή την περίπτωση, και εξετάζουμε και κάποια προγράμματα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και επανεξετάζουμε και όλα τα προγράμματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της βιοπικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να κάνει και μια προσπάθεια εσωτερικού συντονισμού. Νομίζω ότι γνωρίζετε όλη τη σημασία του συντονισμού αυτού, διότι το θέμα των μελισσών δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μία μόνο γενική διεύθυνση. Συμμετέχουν διάφορα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το θέμα των μελισσών και αυτή την άγουσα σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ εγώ κύριε Ντελαντομάντα και να δώσουμε τώρα το λόγο στον εισηγητή Ταμπάτζη για να ολοκληρώσουμε με το θέμα αυτό. Ο... <clears throat> Ευχαριστή συνάδελφοι. Η συζήτηση αυτή κατέδειξε ότι ε, υπάρχουν ε, πολλά έντονα συναισθήματα για το ζήτημα αυτό και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Είδαμε ότι έχουν γίνει, μάλλον ακούστηκε ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικές επιστημονικές έρευνες και πειράματα. Αυτό όμως δεν ισχύει είναι ένα τομέα η μελισσοκομεία όπου δεν υπάρχουν θεμελιώδη δεδομένα. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε καν πόσα μελίσια υπάρχουν, δεν έχουν καταγραφεί. Δεν υπάρχει κανένα καονισμό για τον τομέα αυτό και δεν έχουμε ακριβή αριθμητικά στοιχεία. Κάθε φορά λοιπόν που αναφερόμαστε σε απικίες μελισσών ή σε μελίσια, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας αριθμός συγκεκριμένος, να ξέρουμε για πόσα μελίσια μιλάμε. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές ε, θέσει περιοχές στον τομέα αυτό, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά τα που πάνε ο κύριος Ταραμπέλα και η κυρία Γκαρθία όσον αφορά τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στον τομέα της μελισσοκομείας. Μα ακόμα και για αυτό το ζήτημα δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένη έρευνα στην Ευρώπη. Δεν έχουν τεθεί συγκεκριμένοι ερευνητικοί στόχοι. Αν αναφερθούμε στις μεγάλες εταιρείες παραγωγής γενικά τροποποιημένων οργανισμών, βλέπουμε ότι αυτές δεν θέλουν να δώσουν στους ερευνητές την γενετικά τροποποιημένη εκείνη που θα επέτρεπε να γίνει κάποια έρευνα για την επίπτωση που οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί μπορούν να έχουν στον τομέα της μελισσοκομείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, δεν μπορεί κανεί να λέει αυτή τη στιγμή ούτε ότι έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση, επιζήμια επίπτωση γενικά τροπημένοι οργανισμοί, ούτε το αντίθετο, γιατί απλώ δεν υπάρχουν τα παράτα δεδομένα. Το ίδιο ισχύει και για την έρευνα όσον αφορά τα ζυζανιοκτώνα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζυζανιοκτώνα που ακόμα δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ερευνών για τι επιπτώσει που έχουν στον μιλισσοκομικό τομέα. Σαφώ έχουν γίνει κάποιε έρευνε για κάποια συστατικά, αλλά και πάλι οι έρευνε αυτέ δεν αρκούν και δεν προσελκύουν τελικά το ενδιαφέρον κανενός. Όσον αφορά τώρα τα φαρμακευτικά προϊόντα, δεν υπάρχουν αρκετά τέτοια προϊόντα ακριβώ επειδή δεν υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση εκ μέρους των μελισσοκόμων. Οι μεγάλες λοιπόν εταιρείε παράγουν τα φάρμακα αυτά δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να κάνουν έρευνες να προωθήσουν τα προϊόντα αυτά. Και αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Όπως σας είπα λοιπόν το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιληθεί μόνο αν χρηματοδοτήσουμε την επίλυσή του με κοινοτικού πόρου. Η κυρία Λούλινγκ στη συνέχεια είπε και συμφωνώ μαζί της ότι θα πρέπει απλώς να επαναλαμβάνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει τελευταία 15 χρόνια. Προφανώς δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι ακόμα. Διαφωνώ όμως με τα όσα υπόθηκαν για την κακή οργάνωση του τομέα. Εγώ θα επέμενα περισσότερο στην επιστημονική γνώση που θα έπρεπε να έχουν οι μελισσοκόμοι. Οι ενώσει μελισσοκόμων έχουν συνειδητοποιήσει ότι πολύ συχνά προσπαθούν να θεραπεύσουν τις μέλισσες που ασθενούν με κάποια δικά τους σκευάσματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι μόνο χρηματοδοτικό, υπάρχει και πρόβλημα οργανωτικό αυτή τη στιγμή, πρόβλημα συντονισμού. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Ο κύριος Χάουσλινγκ όπως και άλλοι αναφέρθηκαν στο πρόβλημα αυτό. Και ιδιαίτερα η ξηρασία είναι αυτή που βάλει κατά των μέλισσών. Το ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες χρονικές περίοδοι ξηρασίας, το ότι έχουμε μια υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα φαινόμενα αυτά έχουν σαφώς επιζήμιες επιπτώσεις στην παραγωγή της γύρης και στη μεταφορά της. Διαβάζοντας τώρα την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό μπορώ να πω είναι ότι είναι πολύ καλή. Περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες οι οποίες είναι σε θέση να επιβεβαιώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό, θα πρέπει να συνεχίσουμε την μάχη την οποία ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να, συνεχίσουμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαφορετικά σε 15 χρόνια θα εξακολουθούμε να λέμε τέτοια πράγματα, αλλά ενδεχομένω τότε να μην υπάρχουν πλέον μέλισσες για να σώσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Ταμπάτζη. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 8 μια αποτελεσματική στρατηγική για τις πρώτες ύλες στην Ευρώπη. Συντάκτρια γνωμοδότησης, η Ντατσιάνα Οκτάβια Σάρμπου, επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή, επιτροπή Ήτρε, η κυρία Σαρμπού, η συντάκτρια της γνωμοδότησης, ετοίμασε ένα σχέδιο γνωμοδότησης ε, με το οποίο δέχεται την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη διαδικασία που θέλει να υιοθετήσει, θεωρώντας ότι οι πρώτες ύλε είναι πρωταρχική σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν να δώσουμε το λόγο στη συντάκτρια και να σας υπενθυμίσω ότι επί του θέματος αυτού, το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας, αύριο το πρωί στις 9.30 έχουμε μια σημαντική ακρόαση του καθηγητά Ρεμένο Πρόντι στην Ολομέλεια, στην αίθουσα τη Ολομέλειας. Ε, ελπίζω να μπορέσετε να είστε όλοι παρόντες. Ε, Τατσιάνα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την γνωμοδότηση για μια αποτελεσματική στρατηγική όσον αφορά τα βασικά γεωργικά προϊόντα. Καταρχήν χαιρετίζω την δήλωση, την ανακοίνωση της Επιτροπής, καθώς και την ιδέα να δημιουργηθεί μια στρατηγική ευρωπαϊκή για τα, τις πρώτες ύλες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες ε, προκλήσεις, οι τιμές ε, των ε, πρώτων υλών, αλλά και η αλλαγή των κλιματικών συνθήκων. Ένα φαινόμενο που πραγματικά επηρεάζει την γεωργική παραγωγή και τα αποθέματα παγκοσμίω, τα οποία διαρκώ μειώνονται, ενώ ο πληθυσμό αυξάνεται. Οι τιμές λοιπόν παρουσιάζουν σημαντικέ διακυμάνσει και υπάρχουν και διάφορες ταραχές στην επιστημική αλυσίδα. Χρειαζόμαστε λοιπόν διάφορε δράσει οι οποίες θα μας εγγυηθούν μια συνοχή στην στρατηγική μας όσον αφορά τι βασικές πρώτε ύλε. Μίλησα για τη διακύμανση των τιμών. Όπως ξέρετε, οι αγορές των γεωργικών προϊόντων είναι αντικείμενα πιέσεων. Πρόκειται βεβαίως για μια παραγωγή με εποχιακό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των εισοδημάτων των ε, γεωργών. Χρειαζόμαστε αποθέματα και διαφάνεια, καθώς και πληροφόρηση όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών των πρώτων υλών. Η γεωργία βεβαίως παίζει ένα καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την επιστημιστική ασφάλεια και θα πρέπει να βρούμε τρόπο να καταπολεμήσουμε αυτές τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών. Ελπίζω η νέα κοινή αγροτική πολιτική να συμπεριλάβει κάποια εργαλεία για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Η αύξηση των τιμών δεν μεταφράζεται πάντα με αύξηση του εισοδήματος των γεωργών. Όσον αφορά την κερδοσκοπία, πιστεύω ότι όλες αυτές οι κερδοσκοπικές προσπάθειες θα πρέπει να περιοριστούν. Χαιρετίζω ιδιαίτερα την πρόταση της Επιτροπής να περιοριστεί η εξοχρηματιστριακή δυνατότητα προσφοράς παραγόγων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής, η έκθεση δηλαδή DES θα συζητηθεί αργότερα, σαφώς και είναι ένα καθοριστικό βήμα για να προχωρήσουμε σε περισσότερη ασφάλεια και σε ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τους γεωργούς. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις. Και η τέρμη... Ευχαριστώ Τασιάνο. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 27η Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Ξεκινάει η συζήτηση τώρα. Αν υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο, ο Ζωζέ Μποβέ, ο Αντιπρόεδρος, παρακαλώ. Oui, je... Moi, je salue... Χαιρετίζω την ε, έκθεση αυτή, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστικά συμπληρώνει το όλο σχέδιο μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Νομίζω ότι αυτή τη λογική θα πρέπει να ακολουθήσουμε, να έχουμε δηλαδή μια αποτελεσματική στρατηγική προκειμένου η Ευρώπη να μην εξαρτάται από την διεθνή αγορά γεωργικών βασικών προϊόντων. Ήδη είχε γίνει μια πρώτη συζήτηση όσον αφορά τις φυτικές πρωτεΐνες. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα είχαμε και μία έκθεση όπου λέγαμε ότι ακριβώς θα πρέπει εμείς στα πλαίσια της κοινή γεωρικής πολιτικής να καταφέρουμε να επανακατακτήσουμε και τον τομέα αυτό. Θα δούμε αύριο πώς εξελιχθούν τα πράγματα, θα δούμε πώς εξελιχθεί στο, μέσο, στο μέλλον η κοινή γεωρική πολιτική. Αν καταφέρουμε όμως να συμπεριλάβουμε κάποια σημαντικά βασικά προϊόντα γεωργικά στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής θα εξαρτώμεθα όλο και λιγότερο από τις εισαγωγές των προϊόντων αυτό, αυτών από τρίτες χώρες. Θα εξαρτώμεθα λιγότερο από αγορές όπως η Κίνα και από άλλες αγορές όπως για παράδειγμα στην, από αυτές της Βραζιλίας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια φυτικά προϊόντα με τα οποία τρέφονται τα ζώα, όπως για παράδειγμα η σόγια, η τιμή της οποίας θα αυξηθεί πάρα πολύ και αυτό με τη σειρά του θα έχει επιπτώσεις και στην κτηνοτροφία στην Ευρώπη. Σας δίνω απλώς αυτό το παράδειγμα γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι σήμερα η ε, παραγωγή σε την οτροφική παραγωγή σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει μείωση. Υπάρχει μετεγκατάσταση της παραγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε πραγματικά να διατηρήσουμε μία βιώσιμη παραγωγή στην Ευρώπη, θα πρέπει να καταφέρουμε να διατηρήσουμε βιώσιμο τον τομέα της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε και σε αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Μποβέ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Πολύ καλή ανακοίνωση αλλά και η γνωμοδότηση που έχουμε εδώ. Ενδεχομένως η ανακοίνωση να μην συμπεριλαμβάνονται πολλά στοιχεία όσον αφορά την όλη αλυσίδα παραγωγής και παροχής γεωργικών προϊόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιμείνουμε σε επιμέρους παράγοντες της αλυσίδας που επηρεάζουν τα πράγματα, όπως είπε ο κύριος Ζωζέ Μποβέ για το, το, ζήτημα της σόγιας. Ενδεχομένως λοιπόν μέχρι τις 27 Μαΐου να συμπεριλάβουμε και τέτοια στοιχεία, επιμέρους κρίκους δηλαδή της διατροφικής αλυσίδας στο κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαγκίνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Ποιο είναι εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. My name is ε, Carvalho, Abraham Carvalho. Carvalho ονομάζομαι, προσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι συντονιστής ε, για το ζήτημα αυτό από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και είμαι απο... εργάζομαι, ε, μάλλον εκπροσωπείται αυτή η γενική διεύθυνση ακριβώς επειδή έχουμε να κάνουμε με πρώτες ύλε οι οποίες πολλές φορές χρησιμοποιούνται και στην ε, βιομηχανία. Διαβάσαμε την γνωμοδότηση και θεωρούμε ότι αυτή συνάδει ουσιαστικά με τις απόψεις της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Λέτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια, να γνωρίσετε και εσείς τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με τη διακύμανση των τιμών. Μία παρατήρηση μόνο να κάνω στη φάση αυτή. Στο σημείο 2 αναφέρεστε στον ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων καθώς επίσης και της κερδοσκοπίας όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς απλώς λέμε ότι υπάρχει μια διασύνδεση και λέμε ότι θα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τις εξελίξεις αυτές. Δεν έχουμε καταλήξει λοιπόν εμείς σε μια άμεση διασύνδεση ανάμεσα στη διακύμανση των τιμών και τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι άλλοι που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη διακύμανση των τιμών. Εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές σίγουρα, αλλά και στις ε, αγορές αυτές καθ' αυτές για τα προϊόντα αυτά. Θεωρώ ότι η διασύνδεση αυτή θα μπορούσε να μάλλον υφίσταται, αλλά πρέπει να αναλύσουμε ακόμα περισσότερο πώς οι δύο αυτοί κόσμοι αλληλοεπηρεάζονται. Δεν θα κατέληγα λοιπόν εγώ σε, μια τόσο ξεκάθαρη, σε ένα τόσο ξεκάθαρο συμπέρασμα. Ευχαριστώ. Καλώ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει, να δώσω το λόγο στην Τατσιάνα για να συνοψίσει. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τα σχόλια. Ευχαριστώ και την Επιτροπή. Ελπίζω ότι θα αναλύσετε περισσότερο αυτά που έχω παρουσιάσει και ότι όλα όσα ακούστηκαν θα ληφθούν υπόψη. Molto bene, grazie. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Περνάμε απευθείας στο επόμενο σημείο της διάταξης, πράσινη βίβλος από τις προκλήσεις της ευκαιρίες προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εισηγητής ο κύριος Τζοβάνι Λαβία η ευρωπαϊκή έρευνα θεωρείται ένας από τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης για τη δημιουργία θέσεων εργασία στην Ευρώπη. Ο Τζοβάνι Λαβία ετοίμασε μια γνωμοδότηση που αναφέρεται στην ε, πολλαπλή ε, έρευνα που έχουμε για τον τομέα της γεωργίας και ε, κάνει κάποιες προτάσεις για το επόμενο πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Ε, να δώσουμε το λόγο κατευθείαν στο συντάκτη της γνωμοδότησης και να ζητήσω από τους συναδέλφους να εγγραφούν στον κατάλογο των αγορητών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε γενικές γραμμές είναι πάντα δύσκολο να συνοψίσουμε σε πέντε γραμμές μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας για ένα δύσκολο και διαφορετικό θέμα. Αυτή τη φορά ήταν ακόμα πιο δύσκολο, διότι το να μιλάμε για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι θα πρέπει να σταθούμε σε πολλούς τομείς και να αναλύσουμε πτυχές οι οποίες πόρο απέχουν μεταξύ των θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε φυσικούς πόρους και σε ανθρώπινους πόρους και εκεί επικέντρωσε και την πρόταση γνωμοδότησής μου. Για τους φυσικούς πόρους θεωρώ ότι η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να είναι αυτές οι οποίες θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν ε, τα προβλήματα από την ε, ε, όλο ένα και αυξανόμενη ε, σπάνιδα κάποιων πόρων. Ε, έχουμε όλο ένα και περισσότερο, λιγότερο νερό και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά στο πλαίσιο της συνολικής καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος. Θα πρέπει να προτείνουμε λύσεις για την πιο λογική χρήση των πόρων, είτε βιολογικές είτε φυσικές και επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε οι γεωργικές πρακτικές να είναι πιο παραγωγική και να είναι και το στοιχείο καταπολέμησης της ε, ε, επιδείνωσης του περιβάλλοντος. Όσον αφορά τώρα το ανθρώπινο δυναμικό, θεωρώ ότι είναι στρατηγική σημασία να επενδύσουμε στις δεξιότητες των ανθρώπων μέσω της καινοτομία ε, των υπηρεσιών κατάρτισης, επιμόρφωσης και διαβούλευσης. Θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της ε, επιχειρησιακής δυνατότητας στον γεωργικό τομέα και αυτό είναι σημαντικό για την επιβίωσή τους και επίσης θα πρέπει να τα συσχετίσουμε και με την επιχειρηματική πραγματικότητα. Οι πολιτικές μας θα πρέπει, ιδίω στη γεωργία, να μειώσουν το χάσμα μεταξύ των κόσμων της έρευνας και των κόσμων των επιχειρήσεων και θα πρέπει τα αποτελέσματα να εφαρμοστούν επιτόπου στο χωράφι για να είναι πιο σημαντικές, να είναι στη διάθεση των ε, γεωργικών επιχειρήσεων και από κοινού να βοηθήσουν σε μια πιο καινοτόμα γεωργία προ όφελο και των γεωργών και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Ευχαριστώ όλους όσους θα θελήσουν να συνεισφέρουν στη συζήτηση και να βοηθήσουν να εντάξουμε αυτή την γνωμοδότηση με στοιχεία τα οποία ε, ούτως ή άλλως ε, θα οδηγήσουν στο τελικό αποτέλεσμα με στοιχεία από όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ Τζοβάνι. Η κυρία Πόλσον έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Madame Πόλσον. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον κύριο Λαβία για την πολύ καλή αυτή έκθεση. Όταν αναφερόμαστε στην γεωργία και στις ε, αλλαγές ε, που επέρχονται και που γνωρίζουμε ότι θα λάβουν χώρα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές Καταλαβαίνετε ότι ε, στο κείμενο αυτό βλέπουμε όλες τις ε, προκλήσεις και όλες τις δυσκολίες που εμφανίζονται, αλλά αναφερόμαστε επίσης και σε ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Και θα ήθελα προς αυτό να δώσω δύο παραδείγματα. Πώς δηλαδή μία νέα σύγχρονη γεωργία μπορεί να επιφέρει κάποιες νέες ευκαιρίες μέσω της έρευνας και της εφαρμοσμένης έρευνας. Δεν αναφέρομαι εδώ πέρα μόνο στη βασική έρευνα. Πριν από λίγο αναφερθήκαμε στις μέλισσες, στις μέλισσες μελιτοφόρους, αναφερθήκαμε επίσης σε κάποια επικίνδυνα ζυζάνια, παράσιτα, αναφερθήκαμε επίσης και στις κλιματικές αλλαγές Μιλήσαμε επίσης για κάποιες ε, μεθόδους γεωργίας που φυλακίζουν τον άνθρακα στο έδαφος. Όλα αυτά θα αποτελέσουν πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά της ε, γεωργίας του μέλλοντος. Και θα πρέπει ως προς αυτό να ξέρουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε κάποια φάρμακα, κάποια ζανιοκτώνα, τα οποία θα έχουν δράσει ιδιαίτερα στοχευμένη τα οποία όμως θα πρέπει να χρησιμοποιούν εντελώς επιλεκτικά. Δεν θα πρέπει δηλαδή όπως γίνεται τώρα απλώς να ψεκάζονται τεράστιες γεωργικές εκτάσεις και στη συνέχεια τα φάρμακα αυτά να απορροφώνται από το έδαφος και εκεί πέρα να μολύνουν το περιβάλλον. Αναφερόμαστε λοιπόν στην γεωργία και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει το, τα ύδατα, τους υδατοφόρους υπόγειους ορίζοντες. Ξέρουμε ότι πάρα πολλές φορές η γεωργία, η εντατική βιομηχανική γεωργία καταστρέφει τα θέματα ύδατος. Παράγουμε ουσιαστικά πολύ συχνά τρόφιμα, τα οποία στη συνέχεια στέλνουμε μακριά σε άλλες πόλεις, σε άλλες περιοχές. Φανταστείτε πόσα μέσα μεταφοράς χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή. Φορτηγά, οχήματα, πλοία. Επίσης, δημιουργούνται πάρα πολλά απόβλητα μέσω της α, υφιστάμενης Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές διαστάσεις που υπάρχουν στη γεωργία και σε όλο αυτόν τον κύκλο που δημιουργείται και επιστρέφουμε πάλι στο αρχικό σημείο, πού παράγονται τα τρόφιμα. Βλέπουμε επίσης ότι χρειάζεται να διεξαχθεί έρευνα και σε πάρα πολλούς σημαντικούς τομείς. Για παράδειγμα, η κόκκινη αυτή λάσπη πολλές φορές, η οποία θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί, αφού όμως τύχει κάποιες επεξεργασίες, γιατί περιέχει κάποια συστατικά τα οποία είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Επίσης πάρα πολλές φορές τους αγρούς έχουμε διάφορα φαρμακευτικά υπολείμματα, τα οποία παραμένουν στο έδαφος και έχουν επιζήμιες επιπτώσεις. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα συστήματα αποχέτευσης μέσω των οποίων να καθαρίζονται όλα αυτά τα προϊόντα και να μπορέσουν στη συνέχεια να επαναχρησιμοποιηθούν. Η λάσπη αυτή που περιέχει όλα αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα να καθαρίσει, να καθαριστεί, με συγχωρείτε, και να επαναχρησιμοποιηθεί στις α, γεωργικές εκτάσεις. Ενδεχομένως να μπορεί να είναι ένα πολύ πιο αποτελεσματικό λίπασμα από τα τεχνικά λιπάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε διάφορα προϊόντα. Θα μπορούσε να γράψει κανείς ολόκληρη διατριβή σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν όμως πολλά επιμέρους ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Και νομίζω ένα πολύ σημαντικό μέρος του γεωργικού προπολογισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε έρευνες που επηρεάζουν τελικά την παραγωγή τροφίμων και τη γεωργία. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Πόλσεν. Αν δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο, να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Ρουτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας ε, απευθύνω το λόγο. Είμαι υπεύθυνη για θέματα γεωργίας ε, τροφίμων ε, και τη σχετική έρευνα στην Γενική Διεύθυνση Έρευνας και επιτρέψτε μου να πω ένα-δυο πράγματα εν γέννη για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο και κατόπιν ε, θα σταθώ στις ανάγκε της έρευνας στο γεωργικό τομέα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε αυτή την πράσινη βίβλο για να μπορέσει να λάβει και στοιχεία από όλους τους ενδιαφερομένους και μας ε, χαροποιεί το γεγονός ότι ε, έχετε και εσείς μια γνωμοδότηση. Η δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε ε, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, ε, πολύ ενδιαφερόμενοι έστειλαν στοιχεία, λάβαμε πάνω από 1.300 απαντήσεις από διάφορες πλευρές και επίσης 750 θέσεις από κυβερνήσεις, ε, οργανισμούς και ούτω καθεξής. Πράγματι λοιπόν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και διαθεσιμότητα από τους ενδιαφερομένους να δώσουν τις απόψεις τους και τις ε, σκέψεις τους για το πώς θα πρέπει να συστηθεί το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Και θα υπάρξει και μια διάσκεψη στις 10 Ιουνίου για να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και θα προσκληθούν και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη ε, διάσκεψη αυτή. Και το αποτέλεσμα φυσικά των βασικών σημείων που θα προκύψουν από τη διαβούλευση θα παρουσιαστεί και θα ακολουθήσει και συζήτηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι τρεις βασικοί στόχοι που παρουσιάζονται στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τριπλή. Θα πρέπει να δούμε τις ε, μεγάλες ε, προκλήσεις για την κοινωνία, να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και φυσικά να αυξηθεί η επιστημονική αριστεία και να δοθεί η δυνατότητα να βελτιώσουμε την ερευνητική μας βάση στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημεία τα οποία επεσήμανε και η δική σας επιτροπή στο σχέδιο γνωμοδότησης και ήθελα απλώς να πω ένα-δυο πράγματα για τα σημεία που έχετε αναφέρει εσείς ε, στη γνωμοδότηση και τα σχόλια που ακούσαμε εδώ στη συζήτηση. Όπως γνωρίζουμε, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που μας περιμένει στο μέλλον είναι το πώς θα θρέψουμε τον ολοένα και αυξανόμενο πληθυσμό και γνωρίζετε ότι υπάρχουν προβλέψεις για αύξηση κατά 70% στις ανάγκες τροφίμων τα επόμενα χρόνια Επιπλέον όμως, όπως ε, επισημάθηκε και στη συζήτηση εδώ, υπάρχει και αυξανόμενη ανάγκη και για βιομάζα και για βιοενέργεια και βιοκαύσιμα και αυτό φυσικά προκύπτει από τους ίδιους πόρους. Τα όσα λοιπόν επισημαίνετε εσείς εδώ για την ανάγκη να επικεντρωθούμε στην αποτελεσματικότητα των πόρων και στη σπάνιδα των πόρων όταν αναφερόμαστε στην γεωργική έρευνα, ε, είναι πάρα πολύ εύστοχα. Υπάρχουν ε, κάποιες εκτιμήσεις ε, που έχουμε αυτή τη στιγμή, οι οποίες λένε ότι όχι μόνο χρειαζόμαστε τρόφιμα και καλά τρόφιμα ποιοτικά και σε προσιτές τιμές, αλλά χρειαζόμαστε και περισσότερη βιομάζα για τις βιομηχανίες μας. Για παράδειγμα, η χημική βιομηχανία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή εξαρτάται κυρίως ε, από ορυκτά καύσιμα. Χρησιμοποιούν πετρέλαια και άλλους ορυκτούς πόρους και χρησιμοποιούν μόνο περίπου 8% ε, βιολογικά ανανεώσιμες ε, πρώτες ύλη. Για τους ενδιαφέρει να περάσουν σε πιο ε, βιολογικές πρώτες και αυτές οι πρώτες ύλε θα προκύψουν φυσικά από τη γεωργία και τη δασοπονία. Εάν γίνουν λοιπόν αυτές οι αλλαγές και ε, ο χημικός τομέας και ο τομέας των πρώτων υλών περάσει στην ε, χρήση μια οικονομία που θα βασίζεται στη βιομάζα και αφήσει πίσω του τα ορυκτά, θα έχουμε μια καλύτερη βάση και καλύτερε δυνατότητε καινοτομίε, ώστε να επιτύχουμε δύο στόχου ταυτόχρονα. Να έχουμε επισητιστική ασφάλεια και να καλύψουμε και άλλε ανάγκε, όπω για παράδειγμα τι πρώτε ύλε που χρειάζονται οι βιομηχανίε. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι Υπάρχει μια πολύ σημαντική έρευνα που βασίζεται στην απόδοση, στην σπάνιδα των πόρων και φυσικά ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν και συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα των περιοχών της υπαίθρου και κάποια επιπλέον εισοδήματα φυσικά. Θέλουμε να υποστηρίξουμε και τα όσα είπατε εσείς για την ανάγκη να συνδυάσουμε την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα στη γεωργία και όπως είπατε και εσείς, την ανάγκη να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα θέματα της αλλαγής του κλίματος Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχε οι παρατηρήσει σα και είναι κάποιο από του τομεί του οποίου θα πρέπει να ε, προσέξουμε στον τομέα αυτό. Ο γεωργικός τομέας άλλωστε είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για το μέλλον. Η προσέγγιση που ακολουθήσαμε και επισημαίνουμε το γεγονός ότι η γεωργία είναι ένας από τους τομείς ε, στους οποίους ε, εμφανίζονται οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την κοινωνία, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι συνάδει και με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την κοινοτομία που ζητά να αντιμετωπίσουμε τι μέγιστε προκλήσει στην κοινωνία, ζητούν την αύξηση τη ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα θέλουμε να έχουμε και ένα καλύτερο ε, επιστημονικό πλαίσιο, μια καλύτερη επιστημονική βάση. Και φυσικά ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην ε, μεταβίβαση γνώσεων από τους επιστήμονες στους γεωργούς, είναι ένα από τα σημαντικά σημεία και είναι και μία από τις αδυναμίες που έχουμε διαπιστώσει στο υφιστάμενο σύστημα. Πολλές φορές το καλό επίπεδο γνώσης δεν βγαίνει προς τα έξω και δεν εφαρμόζεται καταλήλως. Μια τελευταία παρατήρηση εδώ για το περιβάλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνδυάσουμε καλύτερα τα πράγματα από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη κατάφερε να αυξήσει την παραγωγικότητά της στη γεωργία. Για παράδειγμα, στην τελευταία δεκαετία καταφέραμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα κατά 20%. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι έχει προκύψει και από την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Τα εδάφη μας έχουν χάσει μεγάλο τμήμα της γονιμότητάς τους, ε, τα είδα τα πλήττονται και επομένως ε, στα επόμενα χρόνια αυτή η κοινή προσέγγιση είναι απαραίτητη για την ε, έρευνα. Πολύ εύστοχη παρατήρηση λοιπόν από πλευρά σας και αυτή. Τώρα, δεν θα ήθελα να κατασπαταλήσω το χρόνο σας. Νομίζω ότι τα σχόλια που έγιναν είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά και περιμένουμε, προσβλέπουμε στην γνωμοδότηση της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ την κυρία Ρουτ, ε, ο Τζοβάνι Λαβία για τις τελικές του σκέψεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο Πόλσεν και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για αυτές τις ε, υποδείξεις και τις συμβουλές. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές συμμεριζόμαστε τα όσα περιλαμβάνει η γνωμοδότηση, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ε, διορθώσεις και κάποιες ε, πιο ε, ειδικέ επισημάνσεις. Συμφωνώ με όσα ακούστηκαν για την αύξηση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο, για την ανάγκη να συνδέσουμε αυτή την αύξηση του πληθυσμού με την παραγωγή διατροφικών προϊόντων, αλλά αυτά δεν θα πρέπει να γίνουν εις βάρος του κοινοτικού περιβάλλοντος. Έχουμε όλο ένα και λιγότερους ε, φυσικούς πόρους, όλο ένα και λιγότερα στοιχεία να χρησιμοποιήσουμε, ιδίω ε, γέες οι οποίες προορίζονται προς τη γεωργική παραγωγή. Θα πρέπει να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα χωρίς να τροποποιήσουμε, χωρίς να αλλάξουμε το περιβάλλον. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε την έρευνα. Πέραν όμως της έρευνας, θα πρέπει να μπορούμε και με τον παραδοσιακό τρόπο, με τη βασική έρευνα, να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση που παράγει η έρευνα στον κόσμο της παραγωγής και στον κόσμο της γεωργίας. Διότι πολύ συχνά δυστυχώς οι καινοτομίε περιορίζονται στα ερευνητικά κέντρα και δεν μπορούμε στην παραγωγική πραγματικότητα να έχουμε την ε, απαραίτητη μεταφορά τεχνογνωσίας που χρειάζεται πραγματικά για να δώσουμε μια νέα όθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας είναι σαφές ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες περαιτέρω προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ λοιπόν για τις ε, χρήσιμες προτάσεις σας ε, και είμαι σε αναμονή των τροπολογιών που θέλετε να καταθέσετε για να βελτιώσουμε την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ Τζοβάνι. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 7η Ιουνίου. Να ευχαριστήσω όλους σας στο σημείο αυτό θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9.30 πριν από τη συνεδρίαση των συντονιστών με τον Υπουργό ε, του Κωσυφοπεδίου θα κάνουμε την ε, συνεδρίαση των συντονιστών ε, στις 5. Στις 5 λοιπόν θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών και 5 και μισή συνεδρίαση με τον Υπουργό του Κωσυφοπεδίου. Ευχαριστώ, τα λέμε αύριο στις 9 και